Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρχίσουμε λοιπόν τη συνεδρίαση μας, αν θέλετε, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Έγκριση μερίσια διάταξης. Έχετε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, μερίσια διάταξη για τη σημερινή και την αυριανή μας συνεδρίαση. Δεν βλέπω. Ωραία. Εγκρίνουμε λοιπόν την μερίσια διάταξη. Πρέπει να εγκρίνουμε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις 23-24 Ιανουαρίου, 6 Φεβρουαρίου, 16 Φεβρουαρίου και 28 Φεβρουαρίου. Όπως γνωρίζετε είναι στο διαδίκτυο τα πρακτικά. Και αν δεν έχει κανένα αντίρρηση, δεν θεωρηθούν ε, εγκεκριμένα μετά το τέλος συνεδρίας. Ανακοινώσεις της Προέδρου δεν έχω σήμερα. Οπότε μπορούμε αμέσω να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η έκθεση του κυρίου Ομαρζέ με θέμα την πρόθεση της συνοχής και της ανάπτυξης σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμογή του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό τον καιρό ετοιμάζει αναθεώρηση της ε, στρατηγικής αυτής του 2012 προς μια εταιρική σχέση για μια ευφυή e ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Το σχέδιο έκθεσης το έχει αναλάβει ο κύριος Ομαρζέ για να γνωμοδοτήσει το Κοινοβούλιο για τη σχέση των περιοχών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα διαμορφωθούν αυτές στο μέλλον. Τώρα θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Ομαρζέ και προτείνω προθεσμή για την κατάθεση των τροπολογιών Δευτέρα 10 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση πρωτοβουλία στο Μάιο. Κύριε Ομαρζέ, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε το σχέδιο έκθεσή σας. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το είπατε κι εσείς. Η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ επίκαιρη και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που αποφάσισε να εκπονήσουμε την έκθεση αυτή. Λέω ότι είναι επίκαιρη γιατί οι παραμονές της εκπόνησης της νέας στρατηγική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανακοίνωση, δεν ξέρω, πάση περιπτώσει ένα καινούριο κείμενο και στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, συζητούμε την έκθεση αυτή. Επίσης, θα διοργανωθεί προσεχώς σε λίγες μέρες και ένα φόρουμ για τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές, πάλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 30 και 31 Μαρτίου. Η παρούσα έκθεση στόχο έχει έναν απολογισμό της υλοποίησης και της εφαρμογής του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες κοινέ πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να κάνουμε λοιπόν όσο γίνεται πιο ακριβή και όσο γίνεται πιο πλήρη την ανάλυση αυτή, εγώ βασίστηκα στην ερμηνεία του άρθρου 349, όπως ε, δόθη το Δεκέμβριο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασε όπως γνωρίζετε στην Ολομέλεια του και επεφάνθη επί του άρθρου 349. Όλοι περιμέναμε ε, την απόφαση αυτή. Θυμίζω περί τίνος πρόκειται στο άρθρο 349. Και το συζητούμε συχνά στην Επιτροπή μας, χωρίς να θυμίζουμε τι ε, ορίζει αυτό το άρθρο. Το άρθρο λοιπόν 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ότι η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών επιδεινώνεται από την απόστασή τους, την απομάκρυνση, την ισιωτικότητα, το μικρό μέγεθος, ε, το ανάγλυφο του εδάφους, τις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες κλπ. Και επειδή πολλές φορές εξαρτώνται από λίγα προϊόντα και στη γεωργική τους παραγωγή. Όλα αυτά μαζί και σε συνδυασμό μεταξύ τους ε, ε, είναι εις βάρος της ανάπτυξης. Το άρθρο αυτό λοιπόν δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να αποφασίζει ειδικά μέτρα για να εφαρμόζονται οι συνθήκε τη περιφέρεια αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερότητε, τι ιδιαίτερε δυσκολίε και προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τα ειδικά προβλήματα αυτά στις διατάξεις της συνθήκης προβλέπουν και τις κοινέ πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, βάσει αυτών των αντικειμενικών συνθήκων αλλά και της νομολογίας θεώρησα ιδιαίτερα εύστοχο για τη δική μας Επιτροπή να ασχοληθούμε επιτέλους με έναν απολογισμό της εφαρμογής του άρθρου 349. Στη συνθήκη του Άμστερνταμ ήταν το 299 παράγραφος 2 Και μετά από 20 έτη εφαρμογής και πλέον και 20 έτη προβληματισμών πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό για το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου. Γράτουμε euh, τις ευκαιρίες ε, της συζήτησης αυτής για να αποτίσω ένα φόρο τιμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δέσμευση, την προσήλωση και τις προσπάθειες που κάνει και ιδιαίτερα η μονάδα, το τμήμα που ασχολείται με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές από την αρχή της θητείας για να κινητοποιήσει και να βιστοποιήσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη να εφαρμόζεται σωστά το άρθρο 349 που έχει και μια διάσταση έτσι εγκάρσια και οριζόντια αδιαμφισβήτητη. Η δική μας Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει ακριβώς αυτές τις αρμοδιότητες τα θέματα που συνδέονται με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Και θα πρέπει να ελέγχουμε σε βάθος, με ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Πάντα στα πλαίσια του δικαίου. Αλλά και στα πλαίσια των πολιτικών προσδοκιών των ενεχομένων στις διάφορες αυτές περιφέρειες. Και εδώ Μιλώ για τις αρχές που ασχολούνται με την περιφερειακή πολιτική αλλά και τους δικαιούχους των ταμείων στις ελόγω Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές διαπιστώσεις που έχετε να κάνει η έκθεση αυτή, η οποία σας έχει διανεμηθεί. Πρώτα απ' όλα υπογραμμίζω ότι μπορεί να υπάρχουν επιτυχίες και συμφωνούμε όλοι σε αυτό, όπως είναι τα προγράμματα POSEI ή με ένα επίδομα για την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους, το άρθρο 349 οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχει πλήρως ακόμα αξιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί. Έχουμε ακόμα λοιπόν περιθώριο ε, και σημαντικό να προοδεύσουμε και στην εφαρμογή του και στην ε, υλοποίηση του. Ιδιαίτερα με συγκεκριμένα προγράμματα ad hoc και νέες ειδικέ ευρωπαϊκές πολιτικές που θα βασίζονται και στα πλεονεκτήματα και στην ιδιαίτερη κατάσταση που γνωρίζουν οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες. Το άρθρο 349, και το λέω χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, έχει ερμηνευτεί και εφαρμοστεί με τρόπο ιδιαίτερα περιοριστικό και δεν έχει επιτρέψει στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες να αναπτυχθούν με βάση τις ανάγκες της ιδιαίτερότητες τους αλλά και τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει εκεί. Άρα είναι εις βάρος των περιφερειών αυτών να εφαρμόζεται με τρόπο περιορισμένο και περιοριστικό αυτό το άρθρο. σε πολλές πολιτικές όπως είναι εμπορική, η θαλάσσια πολιτική, συνοχή, η αλία, η πολιτική ανταγωνισμού ή ακόμα το περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια πολιτική αναπροσαρμογής η οποία ήδη καταλήφθηκε υπέρ ε, μιας ε, ένταξης και προσαρμογής στον κοινό κανονισμό σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες, όπως ας πούμε και την αλληλεία, όπου υπήρχε ένα ποζέι αλληλείας, το οποίο εγκαταλήφθη για την ένταξη ή δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί. Θεωρώ ωστόσο ότι αυτή η διστακτικότητα που υπάρχει που και που από ορισμένε υπηρεσίε να εφαρμόσουν το άρθρο 349 ε, οφείλεται όχι στην κακή θέληση αλλά στην ε, διαθεσμική σύγκρουση ερμηνεών που δίρκεσε σχεδόν 20 χρόνια και που η απόφαση του Δεκεμβρίου 2015 επιτρέπει πλέον να ξεπεραστεί και το σύνολο των θεσμών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Κομισιόν, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο οφείλουν σήμερα να δεχτούν όλα τα, όλες τις συνέπειες και γι' αυτό και παράλληλα με αυτόν τον απολογισμό καλούμε την έναρξη ενός νέου πεδίου στις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές συστάσεις τις οποίες ε, έχουμε περιλάβει σε αυτήν την έκθεση. Ζητάμε αυτό ε, το νέο κεφάλαιο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές να βασίζεται σε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τις εν λόγω περιοχές επί της οποίας εργάζεται η Κομισιόν ε, εκμεταλλευόμενοι πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει αυτό το άρθρο και κυρίως η δημιουργία νέων ειδικών προγραμμάτων και νέων προσαρμοσμένων πολιτικών στις ε, ανάγκες βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης συζητούμε αυτή η νέα στρατηγική να είναι μια στρατηγική σφαιρική και μακροπρόθεσμη που θα δίνει την κοινή προσέγγιση για τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές και που θα συνοδεύεται για κάθε περιφέρεια από στρατηγικό πλαίσιο και συγκεκριμένους στόχους για κάθε μια από αυτές τις περιοχές γιατί βεβαίως υπάρχουν κοινά στοιχεία Γι' αυτό και υπάρχει άλλωστε αυτό το άρθρο. Όμως υπάρχουν ε, επίσης ε, πολλές διαφορές ε, ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές που πρέπει να λεφθούν υπόψη. Επίσης, καλούμε αυτή η νέα στρατηγική να είναι μια στρατηγική πολύ σφαιρική και καλό την Επιτροπή να προβεί την παραμονή της επεξεργασίας αυτής της νέας στρατηγικής ένα συγκεκριμένο απολογισμό της προσέγγισης προς τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές και να εξετάσει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση ε, με λεπτομέρειες για κάθε μια από τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό είναι το, λοιπόν το γενικό πλαίσιο και το έχετε διαπιστώσει κι εσείς η έκθεσή μου στη συνέχεια ε, προβαίνει σε προβληματισμούς ε, πιο συγκεκριμένους μπαίνει περισσότερο στις λεπτομέρειες και εξετάζει πέντε μεγάλους φακέλους κοινοτικής πολιτικής για τους οποίους ε, επίση κάνω κάποιες προτάσεις. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες όλων αυτών των προτάσεων. Θα επανέλθουμε αν το επιθυμείτε στη συζήτηση, αλλά θα σας αναφέρω κάποιες πτυχές που αφορούν πρώτα απ' όλα την πολιτική συνοχή. Για την πολιτική συνοχή θεωρώ ότι Μέχρι στιγμής οι ιδιαίτερα απομακρυσμένε περιοχές λήφθησαν επαρκώ υπόψη, όμως το 349 πρέπει επίσης ε, να ε, ε, παγιωθεί και ιδιαίτερα όσον αφορά τις συνθήκες πρόσβασης στα κονδύλια, τα προγράμματα για την απασχόληση των νέων, καθώς και την πρόσβαση στο σχέδιο Juncker, το ΕΦΣΥ. Τώρα, όσον αφορά την εμπορική πολιτική, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές πολύ σπανίως λαμβάνονται υπόψη και η πολιτική αυτή τελικά εφαρμόζεται χωρίς καμία συνοχή με τους στόχους που έχουν τεθεί σε θέμα τα συνοχής και <clears throat> τους στόχους που έχουμε επίσης θέσει όσον αφορά την γεωργία, στόχους δηλαδή γεωργικούς που θέτουμε σε εφαρμογή στις περιοχές μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλαπλασιάζεται συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών για την μπανάνα, ας πούμε, ή για τη ζάχαρη ε, τους παραγωγικούς τομείς αυτών των ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών που δεν είναι και πολύ άριθμοι και αυτοί, ε, αυτές οι εμπορικέ συμφωνίες πλήττουν τους παραγωγικούς αυτούς τομείς. Γνωρίζετε επίσης ότι με τη μεταρρύθμιση του 2005 οι ποσοστώσεις για τη ζάχαρη και οι εγγυημένες τιμές επίσης καταργήθηκαν. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο όσον αφορά την εμπορική πολιτική που ε, στην ουσία να χαιτίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων αυτών των περιοχών. Αυτό που ζητούμε λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντάξει στις διαπραγματεύσεις και τα συμφέροντα αυτών των περιφερειών ώστε να ε, υπάρξουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες και κάποιες προστατευτικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες. Ο τρίτος τομέας που είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πολιτική της θάλασσας και της αλίας, γιατί γνωρίζετε πως όλες αυτές οι περιφέρειες είναι νησιωτικές περιοχές και υπάρχει και η Γουιάννα με ένα δυναμικό ανάπτυξης στην αλία. Και εδώ επίσης ε, η Ένωση θα πρέπει να συνειδητοποιήσει αυτήν την ε, ναυτική δύναμη την δυναυτική ισχύ που τις προσφέρουν οι απομακρυσμένες αυτές περιφέρειες και θα πρέπει γι' αυτό να προσανατολίσουμε σε αυτό όλα μας τα μέσα ώστε οι πολιτικές αυτές αλλιές να ωφελήσουν κυρίως και πάνω απ' όλα τις εν λόγω περιφέρειες και ο κανονισμός να μην έρθει ακόμα μια φορά να παρεμποδίσει το, δυναμικό, το σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης του τομέα της αλίας στις ε, ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές και η πραγματικότητα είναι ότι ο κανονισμός σήμερα ορθώνει εμπόδια στην ε, ανάπτυξη της αλίας εκεί. Τέταρτος τομέας είναι η φορολογική πολιτική. Ζητώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας των συνθήκων να δεσμευτεί, να εγγυηθεί την παγίωση και την παράταση μετά το 2020 των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που έχουμε εκεί ενισχύει και το επιτρέπουμε και να μην διακυβευτεί έτσι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών από τους εν λόγω κανονισμούς και ε, τα λοιπά. που παραγνωρίζουν και τα αντίστοιχα άρθρα των συνθηκών. Τέλος, διαπιστώνω ότι στην έρευνα, στις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες, στο περιβάλλον, σε όλες αυτές τις πολιτικές, ουσιαστικά ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές, δεν έχουν εκδηλώσει ή δεν έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χωράνε εκεί πολύ σημαντικές βελτιώσεις. Για μας λοιπόν το μέγα ερώτημα είναι το εξής. Να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τα μέσα εκείνα και τα κονδύλια που υπάρχουν σήμερα και υποαπορροφούνται και από τον ορίζοντα 2020. Και εκεί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε ε, τους καλύτερους τρόπους ε, έτσι ώστε να μην μείνουν στο περιθώριο αυτής της μεγάλης πρόκλησης οι περιφέρειας. Μεγάλη πρόκληση εννοώ εδώ την καινοτομία. Και να μπορέσουν και οι τέτρα απομακρυσμένες περιφέρειες να μπουν σε αυτή τη νέα οικονομία της γνώσης. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή θα είναι και πράσινη, όπως η βιοπικιλότητα που έχουν που είναι εξαιρετική και γαλάζια, όπως οι ωκεανοί που ε, τις βρέχουν. Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις ε, παρεμβάσεις και τοποθετήσεις των συναδέλφων για να εμπλουτίσουμε την έκθεση. για τις τροπολογίες περιμένω να τις καταθέσετε και ξέρετε ότι θα φροντίσω να τις ενσωματώσω ειδήσεις όσο γίνεται περισσότερο στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Thank you, thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Μορζέ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και θα δώσω πρώτα τον λόγο στους κοιόδες συζητητές. Κύριε Σκόλτικ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ εκπρόσωπο τον κύριο Πόγκα, ο οποίο απουσιάζει. Και θα μιλήσω στα τσεχικά. Ξεκινώ ευχαριστώντα τον εισηγητή, τον κύριο Μαρζή, για την, το προσχέδιο έκθεση που έχει υποβάλει και για τη συνεργασία που ε, είχαμε και θα έχουμε στην επεξεργασία αυτή τη έκθεση. Θα ήθελα να ανακοινώσει του συναδέλφου ότι ο κύριος Πόγκα συμφωνεί με το σκεπτικό του εισηγητή. Το οποίο σημαίνει ότι ο κύριος Πόγκα και η πολιτική μας ομάδα υποστηρίζει την κατεύθυνση που έχει δώσει στην εκθεσή του κύριος Ομαρζή. Ωστόσο σκοπεύουμε να υποβάλουμε ορισμένες τροπολογίες και θα σας αναφέρω τις κυριότερες από αυτές τις προτεραιότητες μας ε, που θα προσπαθήσουμε να περάσουμε μέσα από τις τροπολογίες. Θέλουμε να τονίσουμε περισσότερο την ανάγκη να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να, υποφελεί, που να ωφελεί τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές της Ένωσης. Επίσης θα θέλαμε να τονιστεί ακόμα περισσότερο στην τελική έκθεση ότι οι περιοχές αυτές έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιαιτερότητες που πρέπει να καλύπτονται από την πολιτική συνοχή και μετά το 2020. Αυτά ήταν τα δύο κυριότερα σημεία που ήθελα να σας μεταφέρω εκ μέρους του κ. Πόγκα. Ο επόμενος ε, σκιώδης ο κ. Μουσκού. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, ξεκινώ συγχαίροντας τον συνάδελφο κύριο Μερζή για το εξαιρετικό προσχέδιο έκθεση που μας έχει υποβάλει. Θα ήθελα όλοι να προσέξουμε και να ε, δούμε ενδελεχώ τα διάφορα προβλήματα που έχει αναδείξει με το έργο του ο κ. Σομαρζή. Τι ιδιαιτερότητε τη αγορά, τον απόκεντρο χαρακτήρα αυτών των περιοχών. Για όλου αυτού του λόγου υπάρχει το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δώσει μια ε, ερμηνεία στο άρθρο 349 ιδιαίτερα ευρεία, κάτι το οποίο επισημαίνει και η έκθεση και το οποίο επιτρέπει να προσαρμόζονται ε, πολλέ πολιτικέ τη Ένωση ε, στο ιδιαίτερο χαρακτήρα των περιοχών μας. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμή δεν έχουν αξιοποιηθεί όπω θα έπρεπε και πλήρω οι διάφορε ε, δυνατότητες που μα δίνει το άρθρο 349 στι πολιτικέ και στα διάφορα προγράμματα η ερμηνεία του μέχρι στιγμής ήταν κάπως περιοριστική και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές είναι πολύ άριθμες το προσχέδιο έκθεσης του κ. Μερζή αναφέρει ότι μια σωστή χρήση του 349 θα μπορούσε να βοηθήσει σε πολλούς τομείς πολιτικής, όπως η αλληλεία, όπως η έρευνα, όπως οι μεταφορές και άλλους τομεί στου οποίους οι από κεντρικέ περιοχές χρειάζονται ακόμα περισσότερη βοήθεια γιατί έχουν πληγεί από την κρίση ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ε, εισαγάγει τον προβληματισμό για το πώς μπορεί να βοηθά αυτές τις περιοχές με τρόπο οριζόντιο, συνολικό σε όλες τις πολιτικές της. Ανταυτού, ε, έχουμε ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις εξοχοσοκέντρες ε, περιοχές και μια αύξηση του αριθμού των εμπορικών συμφωνιών, των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου, το οποίο όμως δημιουργεί κατακαιρματισμό. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε και να δικαιολογήσουμε αυτήν τη ε, διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ της πολιτικής που χρησιμοποιούμε έναντι τρίτων χωρών και ακόμα και περιοχών που είναι μέρη των κρατών μελών της Ένωσης, το οποίο οδηγεί σε προβλήματα οικονομικά για τις περιοχές αυτές και για τους καταναλωτές. Για όλους αυτούς τους λόγους ζητώ να ε, επανέλθουμε και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το 349 της συνθήκης. Αυτό βεβαίως χρειάζεται να ε, ξεκινήσει με ξεκάθαρη πολιτική βούληση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση. Η έκθεση του συναδέλφου ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση κατατείνει και γι' αυτό και την καλυσορίζουμε. Ελπίζω να συνεργαστούμε ε, όλοι έτσι ώστε να υπερψηφιστεί από την Επιτροπή μας και να δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για όλες τις περιοχές της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων και των πιο απομακρυσμένων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Νιούαν. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και τον ε, εισηγητή δεν θα εκπλαγεί βέβαια κανένα συνάδελφος με αυτό που θα πω. Το ECR έχει ορισμένες ανησυχίες για την ειδική μεταχείριση που επιφυλάσσεται στις εξόχως αποκατρισμένες περιοχές εξαιτίας και διά του 349 και ε, είχα την, είχαμε την, την δυνατότητα να συζητήσουμε την θέση του ECR ε, και στο πλαίσιο της συζήτησης που είχαμε σε αυτήν την Επιτροπή για τους στόλους τους αλλιευτικούς. Ο Ίσια θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες ε, που να εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες περιοχές της Ένωσης. Το 349 καλύπτει εννέα συγκεκριμένες περιοχές. Και κατά την άποψη του ΕΣΙΑ αυτή η επιλογή είναι παροχημένη πια. Γιατί υπάρχουν περιοχές, άλλες περιφέρειες στην υπηρετική Ευρώπη, οι οποίες μπορεί να μην είναι γεωγραφικά απομακρυσμένες, οι οποίες μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, αλλά αντιμετωπίζουν και αυτές ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία ε, θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια μεταχείριση αντίστοιχη με αυτή που έχουμε στο 349. Και συμφωνούμε στην σημασία της έκθεσης ε, αξιολόγησης της εφαρμογής, η οποία μας δείχνει ότι ορισμένα από αυτά τα προγράμματα δεν υλοποιήθηκαν ε, ικανοποιητικά. Και θα έπρεπε να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ των κρατών μελών και των απομακρυσμένων, ιδιαίτερως απομακρυσμένων περιοχών. Χρειάζεται να υπάρξουν συγκεκριμένα προγράμματα, στοχευμένα, για την, ε, να βοηθηθούν αυτές οι περιοχές ο εισηγητής σωστά αναφέρει ότι σε διάφορους τομείς πολιτικής, όπως τα γεωργία, η αλία, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν για να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις περιοχές αυτές, τις ιδιότητες απομακρυσμένε και άλλες που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Έχουμε παραδείγματα όπου τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά έχουν επιδείξει ευελιξία. Ένα ως παράδειγμα θα αναφέρω τη σχέση με τη Γουαδελούπη η οποία έχει ένα αριθμό σε χρηματοδότησης 85% ως λιγότερο αναπτυγμένη. Ωστόσο, και, και αυτό παρά το γεγονό μάλλον ότι το, ΑΕΠ ε, αυτών των περιοχών ήταν άνω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν αυτές οι περιοχές δεν ήταν εξόχως απόκεντρες, δεν θα είχαν ιδιαίτερο καθεστώς, ιδιαίτερη βοήθεια. Με την έκθεσή του, ο εισηγητής ζητά περισσότερα προγράμματα πόζη. Και αναφέρει ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρω μέχρι στιγμή. Κατά την άποψη του ECR, η ευέλικτη αντιμετώπιση των απόκεντρων περιοχών υφίσταται παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει α, ε, ακολουθήσει ιδιαίτερα προγράμματα, ιδιαίτερα προγράμματα πόση. Φαίνεται αυτό για παράδειγμα στον τομέα της αλίας. στο ιδιαίτερο ε, στους κανόνες που έχουν επιτραπεί στους αλληλείς αυτών των περιοχών και για την πρόθεση και για την, ε, των προϊόντων τους και για την αλληλεία. Συμπερασματικά, εμείς πιστεύουμε στην ευελιξία, εμείς πιστεύουμε στο ότι χρειάζεται μια υποστήριξη αυτών των περιοχών αλλά αυτή η υποστήριξη θα πρέπει να είναι αναλογική και δίκαιη, έτσι ώστε να μην αδικούνται άλλε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που επίση έχουν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή το 349 αναφέρεται μόνο σε εννέα συγκεκριμένες περιοχές και υπ' αυτήν την έννοια δεν μα επιτρέπει να έχουμε μια δίκαιη αντιμετώπιση όλων των περιοχών που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σμάν Στα γαλλικά, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Μαρζέ για το σχέδιο έκθεσής του, διότι το θέμα αυτό είναι όντως πολύ σημαντικό. Έχω ταξιδέψει κι εγώ λίγο στη ζωή μου και είχα τη χαρά να πάω και στη Μαρτινίκα και στη Ρένιο. Και είναι πολύ μεγαλύτερες οι προκλήσεις από το γεγονός ότι είναι ε, πολύ μακριά από την Ευρώπη. Με τον εισηγητή συμφωνούμε για διάφορα σημεία, ιδιαίτερα για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται τα άρθρα της συνθήκης για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες ε, περιοχές. Επίσης θα πρέπει να διευκολύνουμε και να εμβαθύνουμε τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών αυτών και τρίτων χωρών που ανήκουν ε, στη γεωγραφική τους ε, λεκάνη. Επίσης, θα πρέπει να προβλέψουμε βιώσιμες επενδύσεις, ε, επενδύσεις συγγνώμη, για τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό της γαλάζιας ανάπτυξης που είναι η σε αυτές τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες. Επίσης θέλω να τονίσω την ανάγκη της ε, ενεργειακής αυτονομίας. Ε, είναι πραγματική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, έχουμε και κάποιες διαφωνίες για άλλα σημεία. Πρώτον, έχω μια διαφορετική αντίληψη γενικά σε σχέση με την έκθεση αυτή. Δεν επικεντρωνόμαστε στη συνοχή και την περιφερειακή πολιτική και τι ε, αυτές οι πολιτικές μπορούν να έχουν ως ωφέλη. Ε, στο σχέδιο έκθεσης ακολουθείται μια κάπως μεροληπτική προσέγγιση. Και τι δουλειά έχουν τα εμπορικά ζητήματα. Δεν συμφωνώ καθόλου με τον κριτικό τόνο για τις ε, συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών. Επίσης, διαφωνώ με τη δημιουργία μηχανισμών στήριξης ε, ε, στους παραγωγούς ζαχαροκαλάμου αν πέφτει παγκοσμίω η τιμή τη ζάχαρη. Εμένα μου αρέσει και το ζαχαροκάλαμο και ιδιαίτερα το ρούμι που φτιάχνουν εκεί στη Μαρτινίκα, αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά που πέφτει η τιμή ενό προϊόντο να έχουμε μηχανισμού αντισταθμιστικού ε, αντίθετα στου κανόνε στου οποίου έχουμε συμφωνήσει. Επίση, διαφωνώ με την παράγραφο 35 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Δεν λυπάμαι. Και εκεί διαφωνούμε πάλι, αποκλίνουμε. Ε, δεν λυπάμαι που δεν υπάρχουν κριτήρια γεωγραφικής κατανομής των πόρων στο συγκεκριμένο ταμείο για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένε περιφέρειες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τα διορθωτικά ταμεία που προκρίνουν ε, κάποιες γεωγραφικές ε, ιδιαιτερότητες. Και υπάρχει λόγο γι' αυτό. Είναι διαφορετικά τα ταμεία και λειτουργούμε με διαφορετικό τρόπο. Για όλου αυτού, του λόγους θα κάνω τροπολογίε εγώ στο σχέδιο έκθεση, αλλά βεβαίω ε, είμαι πεπισμένο ότι τελικά η έκθεση θα γνωρίσει μεγάλη υποστήριξη στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και σας κυρία Πρόεδρε. Thank you. Thank you very much, Ευχαριστώ κυρία Presidente. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον συνάδελφο για την έκθεσή του, γιατί πραγματικά χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να δούμε τις πολιτικές επιλογές που θα πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Πρόκειται για περιοχές που δυσκολεύονται λόγω της γεωγραφικής του θέσης, την ε, απομακρυσμένη του θέση, την περιορισμένη έκταση, το κλίμα και η οικονομία τους ε, συχνά εξαρτάται από συγκεκριμένα προϊόντα, γεωργικά συνήθως. Και αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν δέσμευση σε σχέση με την ε, δυνητική του ανάπτυξη. Ακριβώ ο συνάδελφο συζητά ερμηνεία μη περιοριστική του 349 και άρα θετικέ ε, συνθήκε στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών και των γεωργικών προϊόντων. Η αρχή τη αλληλεγγύη είναι οριζόντια και πρέπει να εφαρμόζεται σε όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση ε, σημαντικό είναι το δυναμικό τη γαλάζια ανάπτυξη. Οι θάλασσε οι ωκεανοί αποτελούν κινητήρες της τη τη για την Ευρώπη με τεράστιο δυναμικό για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Η αποκαλούμενη γαλάζια οικονομία απασχολεί 6 ε, εκατομμύρια κόσμο και παράγει ένα δις ε, προστιθέμενη αξία ετησίως. Και οι παράκτης περιοχές της ε, Μεσογείου ωστόσο θα πρέπει να συζητηθούν και άρα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες για συζήτηση για αυτά τα θέματα και άρα συζήτηση για την γαλάζια ανάπτυξη ώστε να πλαισιώσουμε πάντοτε ε, με σεβασμό στα οικοσυστήματα και την διαφορετικότητά του, για να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην απασχόληση, τη βιώσιμη αλληλεία και το σεβασμό της βιοπικιλότητας. Να ξαναρχίσουμε λοιπόν, μάλλον να χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου για τα απόβλητα στην ε, θάλασσα. Ε, 30% μείωση μέχρι το 2020. Αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσει την καινοτομία τόσο στην ε, βιομηχανία της θάλασσας όσο και στην ε, υπηρετική χώρα. Η ναυτική βιομηχανία ρίχνει 80% για την ώρα των αποβλήτων της στη θάλασσα. Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουμε πολλά θέματα. Εάν η προστασία του, του, του, των οικοσυστημάτων αποτύχει, όπως μας ειδοποιούν οι επιστήμονες εδώ και καιρό, όχι μόνο θα βλαφτεί, θα βλαφτεί η, το δυναμικό της γαλάζιας οικονομίας, αλλά ε, θα χάσουμε και τους πόρους ε, και τα όσα κάνουν οι ωκεανοί, δηλαδή τη ρύθμιση του κλίματος και τη σημαντική συμβολή στην ε, βιοπικιλότητα και τη χερσαία. Θα κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις, κάποιες ε, τροπολογίες, αλλά μέχρι στιγμής ε, εκτιμούμε πολύ την εργασία του συναδέλφου Μαρζέ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν ε, το λόγο. Όχι. Τότε θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον Ιστίν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρζέ για την έκθεσή του, η οποία όπως το υπογράμμισε και ο ο ίδιος ε, υπογραμμίζει πριν από το φόρουμ που θα ε, λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα, τονίζει τη δράση της, του συνόλου των βουλευτών ε, από τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές στο Κοινοβούλιο και την οποία δράση χαιρετίζω θερμά. Η έκθεση αυτή βεβαίως προσπαθεί να κάνει ένα απολογισμό για αυτό το περίφημο 349 και είναι βέβαιο ότι μετά από την απόφαση του δικαστηρίου θα ήθελα επίσης να επανέλθω στον τρόπο με τον οποίο μέχρι στιγμής η Κομισιόν έχει εφαρμόσει το εν λόγω άρθρο και πώς το έχει χρησιμοποιήσει. Έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν έχει κάνει προτάσεις, προτάσεις που ήταν απαραίτητες για να ε, ληφθούν μέτρα συγκεκριμένα και που παρατίθενται στην έκθεση σε σχέση με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές επί τη βάση αποκλειστικά του 349 επί διπλής βάσης, δηλαδή τομεακή και 349 ή ακόμα και επί μόνο της τομεακής βάσης, πράγμα το οποίο μας προσάπτει το δικαστήριο στην περιφημή του απόφαση. Όποια και αν είναι όμως η νομική βάση που χρησιμοποιούμε, είτε για θέματα φορολογίας, είτε για θέματα τελωνίας, ε, πολιτικής συνοχής, γεωργίας, ανταγωνισμού, αλληλείας, διεθνούς εμπορίου, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχουν αρκετά και το χαιρετήσατε και εσείς αυτό κυρίο Μαρζή, ότι γίνονται προσπάθειες από πλευρά της Κομισιόν και προτάσεις που έχουν μεταφραστεί σε ουσία. Και αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να εξακολουθήσουμε τη δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι αλήθεια ότι τα μέτρα αυτά τα θυμίζετε στην ε, έκθεση και λέτε πως ε, ίσως να μην ήταν αρκετά ε, αυτό υποστηρίζετε σε αυτό το σχέδιο έκθεσης σας. Βεβαίως και το γνωρίζετε η κυρία η Επίτροπος Κρέτσο που είναι και συντονίστρια στο πλαίσιο της Επιτροπής για τα θέματα των ε, απομακρυσμένων περιφερειών αποδίδει ιδιαίτερο ρόλο ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλήματα των ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών από τους συναδέλφους της. Και αυτό μπορέσαμε να το δούμε ε, στις τελευταίες εμπορικές συμφωνίες, στη δράση της Επιτρόπου Μάλστρομ ε, ή και με τις προσπάθειες της Επιτρόπου Βεστχάγερ στον ανταγωνισμό. Πιστεύω πως εδώ θα είναι θετικός ο απόϊχος και σε πλαίσιο, στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Κομισιόν οι συνάδελφοι προσέχουν όλο και περισσότερο. Μάλιστα σήμερα το πρωί έλαβα μήνυμα από έναν συνάδελφο που μου έλεγε χρειαζόμαστε πιο λεπτομερείς περι... λεπτο... Ε, πληροφορίες για, να διαπραγμα... για τις υπερπεριφερειακές περιοχές για να διαπραγματευτούμε για τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Όλα αυτά πάνε στην καλή κατεύθυνση και πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Αντίθετα, αλήθεια είναι επίσης και το υπογραμμίσατε και εσείς στην εκθεσή σας ότι πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό μάλιστα είναι υποχρέωση που απορρέει από την, ε, το ανακοινωθέν του 2012. Ενώ ταυτόχρονα θα προτείνουμε μια ανανεωμένη στρατηγική για τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Ε, υπάρχει επιθυμία για μια νέα αρχή. Νομίζω και αυτή είναι επιθυμία του Προέδρου της Επιτροπής που το έγραψε. Επιθυμεί μια φιλόδοξη και καινοτόμα ανακοίνωση. Κάποιες φορές νομίζω ότι στην ουσία λέει τα ίδια με την έκθεση, με άλλα λόγια, γιατί λέτε κι εσείς για μια νέα στρατηγική. Τώρα δεν έχω μπροστά μου ακριβώ το κείμενο. Αλλά είναι καινοτόμα και θετική. Ε, αυτό, αυτή είναι η διατύπωση και υπάρχει αυτή η πολιτική ε, βούληση στο ανώτατο επίπεδο της Επιτροπής για στήριξη αυτής της νέας ε, ε, όθησης. Ε, πολλά του έχουν ε, οι, οι για να τα καταφέρουν. Μιλάμε για ιδιαίτερες εξαιρέσεις πάντα, για ιδιαίτερη προστασία, αλλά δεν μιλάμε για τα ατού τους και δεν τις αξιοποιούμε παρκώς. Το έχετε πει και εσείς και οι συναδελφοί σας. Είναι σημαντικό, ε, είτε πρόκειται για την ενέργεια, την κυκλική οικονομία, την γαλάζια οικονομία που αναφέρθηκαν. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουν και αυτά όλα το χώρο τους. Επίσης είναι σημαντικό η, η ΑΠ να υποβάλουν projects μέσα στα οριζόντια προγράμματα και στις πολιτικές και να τις ε, συνοδεύουμε για όλα αυτά Υπάρχουν ήδη projects που αφορούν ε, τις ε, περιφερειακές ε, περιοχές. Η μία έχει, το ένα έχει φτιαχτεί από το, την Γαλλική Υπηρεσία για την ανάπτυξη. Αναπτύσσονται και άλλες πρωτοβουλίες. Πρέπει εκεί να επιμείνουμε και να συνεχίσουμε γιατί θα προκύψουν και άλλα ωραία προγράμματα για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή και πριν τη συζήτηση για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, ε, βεβαίως ε, δεν Ε, ε, θα, ε, θα προηγηθούν και να σας δώσω και κάποιες, κάποια στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Σομαζέ το είπε, την επόμενη εβδομάδα θα λάβει χώρα το φόρουμ για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Είναι σημαντική στιγμή γιατί είναι μια στιγμή που είναι ανοιχτή συζήτηση για το σύνολο των εταίρων και θα αποτελέσει ένα είδος μιας δημόσιας ένα είδος δημόσιας διαβούλευσης για τα θέματα αυτά. Θα είναι η κατάλληλη στιγμή για προτάσεις και συστάσεις που θα μπορέσουν να τροφοδοτήσουν αυτή τη στρατηγική. Αυτή και η συγκεκριμένη έκθεση θα εμπλουτίσει τη συζήτηση αυτή. Και θα συνεχίσει εφόσον κατάλαβα ότι θα υιοθετηθεί τον Ιούνιο. Στόχο είναι να υιοθετηθεί τέλη Σεπτεμβρίου η σχετική στρατηγική, λίγο πριν την σύσκεψη των προέδρων των, των περιοχών ε, των ΙΑΠ που προβλέπεται για τα τέλη του έτους. Να χαιρετήσω και πάλι την εργασία σας. Ε, βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε περαιτέρω ερωτήσεις εάν ε, χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Θα θέλετε να δευτερολογήσετε. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφου που έλαβαν το λόγο και συνεισέφεραν στη συζήτηση που έχουμε σήμερα. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα ε, από τα στοιχεία που ανέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωπος της Επιτροπής. Βεβαίως, ε, συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι πολλά πράγματα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, βεβαίως, και κατά τη διάρκεια της θητείας της ε, σημερινής, της τρέχουσας. Όμως, θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη εφαρμογή του άρθρου 349. Βεβαίως, κανείς δεν αγνοεί, παραγνωρίζει το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ιδιαίτερα προγράμματα υποστήριξης των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών. Και βεβαίω τα γνωρίζουμε αυτά τα προγράμματα, γνωρίζουμε πόσο έχουν υλοποιηθεί μέσω της πολιτικής συνοχής και γνωρίζουμε πόσο έχουν επωφεληθεί και οι περιφέρειες μας. Όμως, όπως είπα και στην αρχή της πρώτης μου παρέμβασης, με την έκθεση αυτή προσπαθούμε να αναδείξουμε το θέμα και έτσι ώστε τελικά όλοι οι επιτροποί να γνωρίσουν καλύτερα ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, αναγνώρισε ότι υπάρχει, ε, μας είπε ότι και ο πρόεδρος Γιούνκερ το αναγνώρισε ότι τίθεται το ζήτημα, στην συνάντηση των ε, προέδρων των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών και το ζήτημα λοιπόν είναι να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Πιστεύω ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο μόνο εφόσον κάνουμε πρώτα έναν απολογισμό του τι συνέβη ως σήμερα, τι καταφέραμε ως σήμερα και επίσης που δεν τα καταφέραμε μέχρι σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάποια θέματα υπήρξαν ε, εμπόδια ή και κάποια τροχοπέδη. Πολλοί συνάδελφοι ορθά επεσήμαναν ότι ιδιαίτερως απομακρυσμένες περιοχές χρειάζεται να επενδύσουν στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Έτσι ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος, να ξεπεράσουμε τα διάφορα προβλήματα μέσω της καινοτιμίας και της έρευνας. Όμως αυτό δεν είναι εφικτό παρά μόνο εάν δοθεί η δυνατότητα στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές να συμμετέχουν στα διάφορα προγράμματα χρηματοδοτικά που κατά καιρούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαιτέρως εκείνα που ανήκουν στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα εμπόδια που τα γνωρίζετε. Ε, τα οποία δεν μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε κονδύλια που χρειαζόμαστε. Γιατί δεν μπορούμε να, συμμετέχουμε, να συμμετάσχουμε σε ορισμένα από αυτά τα προγράμματα ε, εξαιτία περιορισμών. Οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές έχουν και ιδιαίτερα πλέον εκτήματα, ορισμένοι συνάδελφοι τα ανέφεραν. Και πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένε βασικέ στρατηγικέ. Πρώτα απ' όλα, η λεγόμενη κοινή ανάπτυξη και ε, το ζήτημα τη προστασία των ε, ωκεανών. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα, μια καινούργια δραστηριότητα, είναι ένα νέο ε, σύνορο που μπορούμε να διασχίσουμε, η δυνατότητα της εξερεύνησης των κοιτασμάτων που βρίσκονται σε ωκεανούς, ε, το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται η συμμετοχή των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών σε, που βρέχονται από, αυτούς τους, από αυτές τις θάλασσες. Δεύτερη πρόκληση, δεύτερος τομέας προτεραιότητας είναι το θέμα της ενέργειας. Εδώ θα πρέπει να βρούμε συγκεκριμένες ε, λύσεις, γιατί μιλάμε για νησιά Στη Ρεωνιό έχουμε ένα εκατομμύριο κατοίκους. Μικρός αριθμός, αλλά παρόλα αυτά το νησί μας μπορεί να καταφέρει ε, εν ευθέτω χρόνο την ε, ενεργειακή του αυτονομία, αξιοποιώντας τη νεολική ενέργεια, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, μερικές φορές παραγωγή ενέργειας από το υδροηλεκτρική ή ακόμα και τη γεωθερμία. Αξιοποιώντας όλες αυτές τις πηγές ενέργειας θα μπορούσαμε να καταφέρουμε να γίνουμε ενεργειακά αυτόνομοι. Και κάτι αντίστοιχο ισχύει και για άλλες ε, χώρες ΑΚΕ και για άλλα μικρά νησιά του Ειρηνικού. Πρέπει λοιπόν να δούμε πέρα από τα λόγια, πέρα από τις διάφορες χρήσιμες κατά τα άλλα στρατηγικές, να δούμε συγκεκριμένα τι πράττουμε. Ορθά έχει πει ο Πρόεδρος Γιούνκερ ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Επιτροπή της τελευταίας ευκαιρίας για την, για την Ένωση. Ε, κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Αυτή η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνεται ε, για να βελτιωθεί η κατάσταση. Γιατί αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι χειροτέρευση της κατάστασης σε όλες τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Άρα σήμερα πρέπει να κινητοποιηθούμε, σήμερα πρέπει να φροντίσουμε να ξαναέρθουν οι επενδύσεις στα νησιά μας. ετέθη το ζήτημα και εξέφρασαν κάποιοι συνάδελφοι μια αμφιβολία για το κατά πόσον το άρθρο 349 είναι σήμερα ουσιαστικό και μήπω είναι παροχημένο. Το άρθρο αυτό όμως είναι ένα άρθρο της συνθήκης, δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς εύκολα να γνωρίσει. Βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο της ε, νομοθετικής πυραμίδας. Επομένω δεν έχουμε καν δικαίωμα κατά την άποψή μου να ξεκινήσουμε εδώ, σε αυτή την Επιτροπή, μια συζήτηση για το κατά πόσον ήταν σκόπιμο να υφίσταται αυτό το άρθρο. Η συζήτηση αυτή έγινε όταν συμφωνήθηκε η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουμε λοιπόν και πρέπει να το εφαρμόσουμε. Και επενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, θεματοφύλακα των συνθήκων, αυτός ο ρόλος της αποδίδεται, από τη συνθήκη υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα αυτό το άρθρο θα πρέπει να δει το, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πώς θα το εφαρμόσουν εντός του πλαισίου της ερμηνείας του 349 που έκανε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μένα είναι ξεκάθαρο λοιπόν. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την εφαρμογή του 349 ένα άρθρο της συνθήκης. Δεν πάει πιο ψηλά. γιατί αν ορθά κατάλαβα τον συνάδελφο από το ECR, τον κύριο Νιούμαν, ουσιαστικά ζητάτε να αγνοήσουμε το 349. Ή ε, ε, ε, εναλλακτικά να δούμε πώς μπορεί το 349 να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει και άλλες περιοχές. Ναι, σε αυτό το δεύτερο βεβαίως. Μπορούμε να συζητήσουμε για την ανάγκη που υπάρχει να αναγνωριστούν οι ιδιαιτερότητες, ε, οι γεωγραφικές, κλιματολογικές κτλ. και των δικών μας περιοχών, αλλά και άλλων περιοχών, που και εκείνες αντιμετωπίζουν ε, οικονομικά προβλήματα. Προσωπικά πιστεύω στη σημασία που έχουν οι περιφέρειες, περιφερειακές διοικήσεις στην Ευρώπη. Και γενικά ε, δεν πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες με τον ίδιο τρόπο, αγνοώντας το εάν πρόκειται να εφαρμοστούν σε μια περιοχή θαλάσσια, ε, ορεινή, αστική, ε, με πολύ μικρό πληθυσμό, αγροτική κτλ. κτλ. Πρέπει να προσαρμόζουμε τους διάφορους κανόνες, τα διάφορα μέτρα στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, επισημαίνω και πάλι ότι το 349 καλύπτει ε, εννέα συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες έχουν επιπλέον ε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ακριβώς αυτή την, την ιδιαίτερα μεγάλη απόσταση που έχουν από την Ευρώπη. Και γι' αυτό ε, προβλέπονται και ιδιαίτερα μέτρα για αυτές και είναι κάτι το οποίο εξάλλου έχει επιβεβαιώσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην πρόσφατη του απόφαση. Συμφωνώ με άλλους συναδέλφους όπως η κυρία Νταμάτο η οποία αναφέρθηκε στις διάφορων ειδών προκλήσεις και πολιτικές που αντιμετωπίζουμε, στις μεταφορές, στην πολυτροπικότητα κτλ. Ε, για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε σε όλους αυτούς τους τομείς παράλληλα, πιστεύω Ακριβώ, και αυτό λέω με την έκθεσή μου, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα κάνοντα έναν απολογισμό του τι καταφέραμε με βάση το 349 και τα θετικά και τα αρνητικά. για να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάει ακόμα παραπέρα. Στο ζήτημα της εμπορικής πολιτικής, για παράδειγμα, για, το, για τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα πιο αναλυτικά στην ε, συνάντηση ε, με τους σκιώδεις. Εγώ δεν σκοπεύω μέσω της έκθεσής μου να ε, επικρίνω την πολιτική σύναψη συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου με τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αυτό ο στόχος μου. Αυτό όμως που θα ήθελα να αναδείξω είναι πώς μπορούμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα των ιδιαίτερα απόκεντρων περιοχών όταν συνάπτουμε τέτοιες συμφωνίες. Πώς θα φροντίσουμε τα μεγάλα συμφέροντα που συχνά κρύβονται πίσω από τέτοιες συμφωνίες να μην ε, επιβάλλονται στα ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να έχουν οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. και με χαρά διαπιστώνω ότι αυτό αυτός ο τρόπος σκέψης ε, κερδίζει έδαφο εντό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το διαπιστώσαμε στην ε, συμφωνία για τη ζάχαρη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιετνάμ, όπου καταφέραμε τελευταία στιγμή και με δύσκολε διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, συμπεριληφθούν κάποιες εγγυήσει για την παραγωγή ε, ζαχαροκάλαμου από ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. συνεργαζόμενοι με την Επίτροπο Μάλστρομ και μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τη συμφωνία με τον Ισημερινό, όπου τελευταία στιγμή και πάλι συμπεριελήφθηκαν συγκεκριμένες εγγυήσεις στη συμφωνία και ένας μηχανισμός προστασία, μια ρήτρα προστασία. Και παρεπιπτόντω θα ήθελα για αυτό το θέμα να ευχαριστήσω και την ε, ομάδα Άλντε ε, για τον πολύ επικοδομητικό ρόλο που έπαιξαν ε, στο να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία. Έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα και πιστεύω ότι πλέον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι εκ των προτέρων απριόρι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα συμφέροντα και οι ανάγκες των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών όταν ξεκινάμε διαπραγματεύσεις ε, για τη σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας. Αυτά από την πλευρά μου κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και ε, με μεγάλη ε, χαρά θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους, περιμένω τις τροπολογίες που θα υποβάλουν στόχος μου είναι να καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα υπερψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή μας και μετά στην Ολομέλεια για να βοηθήσουμε αυτές τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θυμίζω την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Τη Δευτέρα 10 Απριλίου είπαμε στις 12 το μεσημέρι. Για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας το Μάιο. Oh. Uh, λοιπόν, ένα διάλειμμα 15 λεπτών τώρα είναι ότι πρέπει για καφέ, γιατί περιμένουμε τον ε, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κατάινεν, στις 4.30.

Ladies and gentlemen, dear colleagues, may I ask you to take your seat. Παρακαλώ, καθίστε για να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Με το επόμενο σημείο στην ημερήσια μας διάταξη, όπου έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε σήμερα τον κύριο Γιούρκη Κατάινεν, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής που είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη, την απασχόληση, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Σήμερα θα συζητήσουμε την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την παράταση αυτού καθώς και να τεχνικά να βελτιώσουμε και το Ταμείο αλλά και το Ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα. Επίσης ε, θα τον ρωτήσουμε τη γνώμη του για την συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο τα Ταμεία και το ΕΦΣΥ και βεβαίως απαντήσεις σε ερωτήσεις ε, από πλευράς των μελών. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων αποτελεί τμήμα τη συνεχιζόμενη εργασία ε, ελέγχου τη Επιτροπής και με χαρά θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήσεις, ε, αρχίζοντας με τους συντονιστέ των πολιτικών ομάδων. Έχετε το λόγο κυρία Κατάινεν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Σα ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε το μέλλον του ΕΦΣΥ το πώς έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα και πώς και θα θέλαμε να το αλλάξουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το ΕΦΣΥ θα παίξει το ρόλο του στην προώθηση της ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη. Το ΕΦΣΥ λοιπόν λειτουργεί εδώ και 1,5 χρόνο και φαίνεται να λειτουργεί αρκετά καλά. Έχουμε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα 28 κράτη-μέλη για 32 δις περίπου. Συγχρηματοδότηση σημαίνει δάνεια ε, για έργα υποδομών ή για βιομηχανικές επενδύσεις ή με σο τραπεζών ε, προς τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, αυτά τα 32 δις εγγύησεις, ευρωπαϊκές εγγύησεις θα κινητοποιήσουν γύρω στα 170 δις που πανεπενδύονται. Δηλαδή 32 δις από το ΕΦΣΥ μοχλεύουν πραγματικές επενδύσεις αξίας 170 δις. Είναι λίγο περισσότερο από το ίμιση του στόχου μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για τη χρηματοδότηση των ε, μικρομεσαίων που είναι επιτυχές. Όπως είπα, το ΕΦΣΥ χρηματοδοτεί και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω τραπεζών, δηλαδή τραπεζών που λειτουργούν στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες ή ενδιαμέσως μπορεί να είναι επίσης μια εθνική τράπεζα ή κάποιο επισφαλές κεφάλαιο ή κάποιο επενδυτικό ταμείο. Έχουμε λοιπόν αυτή την, ε, τον, τον συνδυασμό και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που υποστηρίζεται και στα κράτη-μέλη. Και έχουμε έτσι παροχή χρηματοδότηση σε περίπου 400.000 μικρομεσαίες στην Ευρώπη. Χάρη σε αυτές τις συμφωνίες λοιπόν, 400.000 μικρομεσαίες θα χρηματοδοτηθούν. Και γι' αυτό τον λόγο και αποφασίσαμε να χορηγήσουμε περισσότερους πόρους στο ΕΦΣΙ και στις μικρομεσαίες. Γιατί το πρόβλημα για τις, για τις μικρομεσαίες είναι η χρηματοδότηση σχεδόν παντού στην, στην ε, Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα την γεωγραφική κατανομή, Το ΕΦΣΙ ε, είναι ένα πρόγραμμα που δεν έχει να κάνει με τη γεωγραφική κατανομία. Αλλά ε, ωστόσο φαίνεται να υπάρχει και μια αρκετά ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή. Να σας δώσω ένα κατάλογο με δικαιούχους. Η Εστονία είναι η πρώτη. Αν δούμε δηλαδή τον αντίκτυπο του ΕΦΣΙ ΑΕΠΑ. Η Βουλγαρία δεύτερη, μετά η Ισπανία, μετά η Λιθουανία μετά η Πορτογαλία, έκτη η Ιταλία, έβδομη η Ελλάδα. Και μετά είναι άλλες χώρες. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε για αυτό το θέμα της γεωγραφικής κατανομής, γιατί υπάρχουν χώρες όπως για παράδειγμα η Ρουμανία, που δεν έχει ωφεληθεί τόσο από το Εύση... η Μάλτα, η Κύπρος, Επισκέφτηκα την Ρουμανία όπως επισκέπτομαι όλα τα κρατημέλη, αλλά αν για παράδειγμα συγκρίνουμε τη Βουλγαρία με τη Βουλγαρία, δεν ξέρω πόσο είναι δίκαιο να τις ε, συγκρίνουμε, πάντως είναι γειτονικέ χώρες τουλάχιστον. Στη Βουλγαρία ήδη έχουμε τρεις συμφωνίες για χρηματοδότηση μικρομεσαίων, συν ένα-δύο άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΦΣΥ. Ενώ στην Ρουμανία καμία τράπεζα δεν ε, δήλωσε προθυμία για να χρησιμοποιήσει το εύση για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όταν τελευταία μου επίσκεψη στη Ρουμανία ρώτησα τους τέσσερις διοικητές των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών, είπαν ότι δεν υπάρχει ζήτηση για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων στη Ρουμανία. Εγώ βεβαίως πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό, γιατί αν συνέβαινε αυτό η Ρουμανία θα ήταν η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου δεν χρειάζεται χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες. Εν πάση περιπτώσει, για κάποιο λόγο ε, αυτή είναι η αίσθηση, ότι δεν υπάρχει ανάγκη. Πάντως πρέπει να περάσουμε και να προσέξουμε τη γεωγραφική κατανομή και οι τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναβαθμίσει την παρουσία της επιτόπου, δηλαδή έχει περισσότερους ανθρώπινους πόρους τοποθετήσει στα τοπικά γραφεία, στα κράτη-μέλη και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την τεχνική αρρωγή και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις χώρες συνοχής. Διότι κάποιες φορές, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από ότι εγώ, οι αρχές δεν έχουν πάντα τις απαραίτητες δυνατότητες για να ε, συστήσουν προγράμματα ναι, ε, ή όταν ε, βλέπουμε άλλες ευκαιρίες, δηλαδή συνδυασμό με άλλα κονδύλια από την Ένωση και το ΕΦΣΥ, για παράδειγμα τα διευθυντικά ταμεία ή την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, που μπορούν ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσουν μαζί με το ΕΦΣΥ. Δεν έχουμε την πρόθεση να ανακατανύμουμε πόρους από τα διαφορετικά ταμεία στο ΕΦΣΙ. Απλώς θέλουμε να καταστήσουμε ευκολότερη ευκολότερο το συνδυασμό διαφορετικών χρηματοδοτικών πόρων ε, με το ΕΦΣΙ. Αυτό ήταν ο στόχο ε, του αναθεωρημένου κανονισμού. Οι τοπικέ, περιφερειακέ και εθνικέ αρχέ να μπορούν πιο εύκολα να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα διαρθωτικό ταμείο και εύση, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν και ιδιωτικού πόρου που υπάρχουν ήδη στην αγορά. Οπότε, εξαρτάται από τους ίδιους τους δικαιούχους ε, αν θέλουν να συνδυάσουν διάφορα μέσα χρηματοδοτικά της Ένωσης ή όχι. Μια βασική αξία του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων είναι ακριβώς η ε, παροχή και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα όσα πράττει κατά κανόνα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μέχρι τώρα έχει λειτουργήσει αρκετά καλά αυτό, αλλά θέλουμε στο μέλλον να ε, γίνει ακόμα καλύτερα. Τμήμα λοιπόν της, πρόθεσης, της προτείνουμε για το FC2 όλες οι επενδυτικές αποφάσεις να τεκμηριώνται και να εξηγούνται δημοσίως. Για ποιο λόγο επελέγει το συγκεκριμένο έργο και πού είναι η προστιθέμενη αξία κάθε φορά. Ε, first of all, FC. Καταρχά, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν θα πρέπει να κάνει ακριβώ τα ίδια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και δεύτερον, δεν θα πρέπει να ε, ε, εξωθεί από την αγορά τις ιδιωτικές ε, επενδύσεις. Στόχος δεν είναι να διώξουμε τους ιδιώτες από την αγορά. Το αντίθετο είναι να συγκεντρώσουμε για σδίτ ιδιώτες. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω θα σταματήσω εδώ ε, διότι ε, θέλω να αφήσω όσο γίνεται περισσότερο χρόνο στα μέλη για ερωτήσεις και για σχόλια. Εμείς τις δικές σας απόψεις θέλουμε να ακούσουμε και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω ε, όσο μπορώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Αρχίζουμε λοιπόν με τις ερωτήσεις. Οι συντονιστές. Πρώτη, ο κύριος Νοβάκοφ ο κύριος Νοβάκοφ είναι ο νέος συντονίστης. Ναι. Όχι, όχι, ας πούμε είμαι μιλητής προς το παρόν. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ομιλία σας και για την παρουσία σας εδώ. Σήμερα δεν χωρά καμία αμφιβολία. Είναι πάντα θετικό και γόνιμο να έχουμε την ευκαιρία να συζητούμε μας ε, εξηγήσατε ποιες είναι οι προθέσεις σας και οι στόχοι σας με την ε, νομοθεσία Omnibus που είναι από τα σημαντικότερα νομοθετήματα των τελευταίων πολλών ετών. Πραγματικά εστιάζεται στην προσέγγισή σας. Επανειλημμένα αναφέρετε τις συνέργειες μεταξύ του το Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, συνδέοντας την Ευρώπη, το Κοινωνικό Ταμείο κτλ οι συνέργειες αυτές δεν είναι μόνο εφικτές, αλλά ενθαρρύνεται και όλό τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να προσπαθούν να συνδυάζουν διαφόρους ε, πόρους χρηματοδοτικούς και διάφορα ταμεία. Εδώ υπάρχουν ε, μερικά εμπόδια για το συνδυασμό διαφόρων οικονομικών πόρων και χρηματοδοτικών ε, όπως είναι η νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις. Παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν ε, θα πρέπει να καλύπτει ή να καλύπτεται μάλλον από, το ταμείο, από, από την νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις ενώ άλλα ταμεία υπάγονται. Ε, και όταν έχει συγχρηματοδότηση από διάφορα ταμεία, τι γίνεται. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε. Γιατί οι συνάδελφοί μου ταξιδεύουν πολύ, πηγαίνουν σε εκλογικέ του περιφέρειες και προσπαθούν να εξηγήσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση πώς θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν περισσότερο από εσά. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρέα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Κατάινεν. Ξέρετε ότι είμαι συγγήτρια για τη διαδικασία Omnibus, την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και για να είμαι ειλικρινής, αν ε, συνδέσουμε το, ε- ή συγκρίνουμε το ΕΦΣΙ με το ΕΖΙΦ και θέλουμε να έχουμε και συνέργειες, ε, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το ΕΦΣΙ έχει τελείως διαφορετική στόχευση από τα ταμεία ΕΖΙΦ που είναι κυρίως για την περιφερειακή, κοινωνική και οικονομική συνοχή. Το ΕΦΣΙ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, είναι κάτι ε, που διαθέτει δημοσίους πόρους για να προσελκύσει ακόμα περισσότερους ιδιωτικούς με λίγα κριτήρια, αλλά δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση όλα αυτά με την πολιτική συνοχή. Αυτό λοιπόν είναι ένα τμήμα της δυσκολίας, αν θέλουμε να το συνδυάσουμε με τα ταμεία έζη. Καταρχήν λοιπόν για μένα έχει νόημα, το θέλουν τα κράτη-μέλη. Όταν θέλουν να κάνουν έργα στην πολιτική συνοχή, να τα χρηματοδοτούν από το ΕΦΣΥ. Υπάρχει αυτό το εργαλείο, αλλά είναι πάρα πολύ περίπλοκο και στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να εφαρμόζεται. Γι' αυτό είναι σχετικά λίγα τα κράτη-μέλη που το έχουν πράξει. Και μάλιστα διαμαρτύρονται κιόλα και κάνουν παράπονο ότι είναι πολύ περίπλοκο. Και έκανε μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία επεξεργαζόμαστε, για να εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα με κάποιε προποθέσει και κάποια κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται και να τηρούνται για να απλουστευτεί όσο γίνεται. Υπάρχουν εκεί πολλές δυνατότητες να συμφωνήσουμε και περιθώρια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί όμως που έχω εγώ πολύ μεγάλες επιφυλάξεις είναι ο συνδυασμός των προτινόμενων ε, ταμείων. Αυτό που μας είπατε από τα διαρθρωτικά ταμεία και από τα ταμεία ΕΣΥΦ να αντλούν πόρους στα κράτη-μέλη και με δική του ε, συνεισφορά, ε, πάντα εθελοντική, να τα επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, την κεντρική διαχείριση. Και η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχωράει τόσο πολύ που ορίζει κάποια πραγμάτα που δεν έχουν αποφασιστεί ούτε στο ΕΦΣΙ, όπως είναι η πρώτη απώλεια, first loss. Αυτά είναι θέματα συναπόφασης. Και δεν είναι δυνατό να τα αποφασίζουμε ή να τα περαιώνουμε εδώ και τώρα. Αφήστε που δεν συμφωνώ και δεν το εγκρίνω. Όταν πρόκειται για χρήματα, όποια και να είναι αυτά, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης και χωρίς δυνατότητα να υπάρχουν κάποια κριτήρια να επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να εξηγεί που τα δίνει. Ξέρω ότι υπάρχουν φόβοι ε, να μην ε, μπορεί μια χώρα να απορροφήσει 10 δισεκατομμύρια ή 15 δισεκατομμύρια ε, ευρώ από τα ταμεία ΕΣΥΦ και να τα επιστρέφουν στους υπουργού οικονομικών των κρατών μελών, του κάστοτε κράτους. Κανείς δεν το θέλει αυτό στην Επιτροπή μας ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι διαχείρισης. Θα παρακαλούσα λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλει να εμείνει σε αυτή την πρόταση, να φέρει νέα πρόταση και όταν ε, έχει έρθει ο κανονισμός fc 2.0, και γνωρίζουμε τι έχει πει ο νομοθέτης ή οι δύο συνομοθέτες για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να δούμε αν είναι δυνατός αυτός ο συνδυασμός με ποιες προϋποθέσεις και ποιους όρους, με ποιες διαδικασίες, πώς μπορεί κανείς να τις επιλέξει κτλ. Και ποια θα είναι η συμμετοχή στα κράτη-μέλη και με ποιο τρόπο αυτή θα οργανώνεται. Όλα αυτά δεν είναι εύκολες αποφάσεις. Θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια ότι είχαμε προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη με το κοινωνικό ταμείο, ότι το είχε υποαπορρόφηση. Αυτά έκτοτε άλλαξαν, αλλά υπήρχαν κάποιες κυβερνήσεις τότε κρατών μελών που ζητούσαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν ε, χρήματα από το Κοινωνικό Ταμείο και να συνδυάσουν τους πόρους με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΦΕΝΤΕΡ. Καλό ήταν που ήταν τα κριτήρια έτσι πιο αυστηρά για να μην κάνουν ό,τι θέλουν τα κράτη-μέλη, αλλά επαναλαμβάνω και με χαρά να το επαναλάβω όσο χρειάζεται. Η πολιτική συνοχής είναι ένα σημαντικό εργαλείο ακριβώς σε καιρούς όπου ακούμε πολύ κριτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί αυτό το μέσο να δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτικούς στόχους που υλοποιεί ε, μαζί με πολίτες επιτόπου στην περιφέρεια και αυτά είναι ορατά, χειροπιαστά. Καταλαβαίνει ο κόσμος και βλέπει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δική τους ζωή, πώς μπορεί να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν και τους βοηθάει να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους. Και εδώ είναι μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αν τη ε, διαχείριση είναι ε, όσο γίνεται πιο αποτελεσματική και πιο διαφανής. Και δεν με βοηθάνε οι μεγάλες εκστρατείες που κάνετε για να επιστρέφουμε χρήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που με βοηθάει είναι να βελτιωθούν οι διαδικασίες και να απορροφούνται τα κονδύλια στην περιφέρεια. Για τη συγκεκριμένη πρόταση λοιπόν, της προ... Ε, το συγκεκριμένο τμήμα της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη δική μου υποστήριξη δεν πρόκειται να την έχετε. Και επειδή βλέπω και τις τροπολογίες των συναδέλφων, είναι μεγάλη η πλειοψηφία στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, και αντίστοιχα θα ισχύσουν και στην Ολομέλεια. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει και να μην εμείνει να το επιβάλλει αυτό με τον οποιοδήποτε τρόπο. Δεν πρόκειται να βοηθήσει. Είναι τελέσφορο κάτι τέτοιο. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Κύριος Νιούμαν. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Με χαρά το ECR διαπιστώνει ότι σε διάφορους τομείς η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρει να ανακάμψει από την οικονομική κρίση, ωστόσο συνεχίζουν ε, πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα η ανεργία και το γεγονό ότι στου ε, μακροχρόνια ανέργου το ποσοστό τη ανεργία είναι διπλάσιο από αυτό το, που είχαμε το 2008. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ε, έλλειψη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση του προβλήματο αυτού, ιδιαίτερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, θα, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν καλωσορίζουμε προγράμματα τα οποία ε, απευθύνονται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί χρειάζεται να αυξηθεί ο αριθμός των απασχολούμενων σε αυτές και να ξεφύγουμε από τη στασιμότητα. Όπως γνωρίζετε, το 16% του διαθέσιμου κεφαλαίου ήταν, προερχόταν από, την, από το Ηνωμένο Βασίλειο και 7 έως 8% των επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του 2015 ε, από την Τράπεζα Επενδύσεων κατευθυνόταν προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποιο, πώς βλέπετε τις, προ, τις προοπτικές σε σχέση με όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Ε, σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είχαμε και παλαιότερα την ευκαιρία να συζητήσουμε για το σχέδιο Juncker. Το ονομάζω σχέδιο Juncker γιατί βεβαίως υπάρχουν και εκείνοι που μας παρακολουθούν από το ίντερνετ και με τα κρονίμια ΕΦΣΙ ίσως να μην μας καταλαβαίνουν. Γνωρίζουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Ε, ας μιλάμε για το σχέδιο Juncker που είναι ξεκάθαρο. Από τη δική μου την πλευρά δεν έβρισκα κανένα λόγο να αντιταχθώ σε ένα πρόγραμμα, στο πρόγραμμα αυτό, που προσπαθεί να δημιουργήσει ε, ανάπτυξη και να ε, κινητοποιήσει και πάλι τις επενδύσεις. Στοιχείο κρίσιμο, στοιχείο κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος είναι το πόσο γρήγορα θα μπορέσει να ανταποκρίνεται στις αλλαγές. Και όπως γνωρίζετε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε προσυλλομένοι σε ζητήματα αρχών, σε ζητήματα κανονισμού, σε διαδικασίες και είναι λογικό. Ωστόσο, θα ήθελα να προσέξουμε όλοι, να μην πέσουμε στην παγίδα εξαιτία αυτού του, ε, της, της ε, στους τύπους να, χάσουμε, να, να οδηγήσει στο να μην έχουμε την ταχύτητα ανταπόκρισης που χρειάζεται Δεύτερον, η Επιτροπή Περιοφυρικής Ανάπτυξης ανησυχούσε από την αρχή, το οποίο είναι λογικό και συνεχίζει να ε, το θεωρεί αυτό προτεραιότητα, να μην δημιουργηθούν προβλήματα στα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης, τα περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ που βρίσκονται στα ταμεία αυτά. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να συμπεριληφθούν στον τρόπο με τον οποίο θα αποδίδονται οι χρηματοδοτήσει από το πρόγραμμα Juncker γεωγραφικά κριτήρια, κριτήρια γεωγραφική ισορροπία. Το ερώτημα μου θα ήταν το εξή, αν θα μπορούσατε να δώσετε στην Επιτροπή μας μια φωτογραφία της κατάστασης σήμερα, πώς έχουν κατανεμηθεί τα διάφορα κονδύλια. ακολουθώντας ε, τις ε, διάφορες ε, κατανομές των περιφερειών σε μικρότερες, μεγαλύτερες, αναπτυγμένες, λιγότερο αναπτυγμένες κτλ. Έτσι ώστε να γνωρίζουμε τελικά πόσα ήταν τα χρήματα που κατευθύνθηκαν προς περιοχές σε λιγότερο αναπτυγμένες και πόσα σε περισσότερο αναπτυγμένες. Νομίζω χρήσιμο θα ήταν να τα γνωρίζουμε αυτά, τα στοιχεία, Ίσως θα διασκεδάσουν και ορισμένε από τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι συνάδελφοι. Ελπίζω τουλάχιστον, αν δεν μπορείτε να μου απαντήσετε αμέσως, στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για τα κριτήρια γεωγραφικής ισορροπίας που ακολουθεί. Και έρχομαι στο τρίτο θέμα που είναι η τεχνική βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό να, είναι, να γίνει γνωστό σε όλους ότι υπάρχει διαθέσιμη τεχνική βοήθεια η οποία μπορεί να δοθεί σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, Εκριβώς σε εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στις εθνικές αρχές για να τους ε, βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ κύριε Ντεμάτου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως πάντα και σήμερα έχω την εντύπωση ότι ακούμε ωραία λόγια πολύ ε, ελκυστικές υποσχέσεις, αλλά είναι πάντα οι ίδιες. Από τότε που πριν από 1,5 χρόνο υποβλήθηκε αυτό το σχέδιο που έπρεπε να εγγυηθεί η προσθετικότητα, στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και που υποσχόταν να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Στη διάρκεια της παρουσίασης του Λευκού Βιβλίου για την Ευρώπη ακούσαμε και τον πρόεδρο Γιούνκερ να λέει πως η Ευρώπη Μα δεν είναι αυτή που θα εγγυηθεί για, τις, για την απασχόληση, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε. Από ένα από τα δύο θα γίνει. Τώρα για το ΕΦΣΙ έχουμε ακόμα και πολλές αμφιβολίες. Παρενέβη το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο που έδειξε την ε, πιθανή στασιμότητα του εφέ μοχλού ε, ένα εφέ μοχλού το οποίο πάντοτε υπολογίζεται μοιράζοντας, διαιρώντας μάλλον ε, το τελικό αποτέλεσμα ενός έργου ε, με το ποσοστό που συμβάλλει το εύση. Είμαστε βέβαιοι όμως ότι αυτά τα έργα θα έχουν αίσιο πέρας. Από την πύρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ε, μεγάλη αύξηση των έμεσων ε, χρηματοδοτήσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως είναι εξαιρετικά αδιαφανής η δομή και υπάρχουν ε, διάφορες κερδοσκοπικές κινήσεις με στόχο τη μεγιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων κερδών παρά την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το ΕΦΣΙ και το ΕΦΕ μόχλευσης δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως ε, παραβάν για να καταπιούμε πιο εύκολα το χάπι της παράτασής του. Κύριε Κατάιναν, είπατε ότι είστε πάντα διαθέσιμος να συζητήσετε μαζί μας, αλλά θέλω μια παραπάνω προσπάθεια να καταβάλλετε. Να κάνετε δηλαδή κάποιες απαντήσεις να δώσετε μάλλον για το ΕΦΣΙ, αλλά και για την ΕΤΕΠ. E Τι είδους ε, ε, ανάπτυξη θέλουμε. Εν γέννη ακούμε για βιώσιμη ανάπτυξη. Όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα στηρίζονται ε, τα, τα στερεά καύσιμα, ε, τα ορυκτά καύσιμα. Ακόμα στηρίζονται λύσεις ε, στηρίζονται λύσεις οι οποίες ρηπαίνουν, όπως στο Τάραντο. Έχετε εκτιμήσει τον αντίκτυπο των διαφόρων προγραμμάτων που στηρίζετε ε, και την προστιθέμενη αξία του κάθε έργου και πώς αυτό μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων του ΕΦΣΥ για να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε επίσης να έχουμε και γραπτός μετά από αυτή τη συνεδρίαση τα στατιστικά στοιχεία τα απομαδοπαϊμένα σε σχέση με κάθε project που χρηματοδοτείται και τα δάνεια που δίνονται μέσω του ΕΦΣΥ, μέσω των ε, διαφόρων ενδιαμέσων, τις ε, αξιολογήσεις ε, εξάντε, εξπόστη για κάθε project με συγκεκριμένους δείκτες και κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, η Κομισιόν θα μπορούσε να μας δώσει τουλάχιστον κάποιες διαφανείς ενδείξεις για το πόσα χρήματα δίνονται στους ενδιάμεσους χρηματοδότες και πόσο πραγματικά φτάνει στους τελικούς δικαιούχους για κάθε ένα project. Περιμένω την απάντησή σας και σας ευχαριστώ. Thank you. I have... Uh, ευχαριστώ. Έχω πολλούς ακόμα. Έξι περίπου συναδέλφους, τους εξής επτά. να ομαδοποιήσουμε όλες τις ερωτήσεις και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κατάινεν. Κυρία Βέστιφα, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί με κάλυψε η συνάδελφος Κρέλ. Ε, μίλησε πολύ για τις αγωνίες και τους φόβους. Είμαι και εγώ εισηγήτρια, έχω διατελέσει για την αστική ανάπτυξη, για το θεματολόγιο των πόλεων και αύριο θα παρουσιάσω την έκθεσή μου για τη μελλοντική πολιτική συνοχή. Η κυρία Κρέλ πραγματικά ανέφερε αυτά που με απασχολούν και μένα με τρόπο πολύ ξεκάθαρο. Θα ήθελα να σας επιζήσω την προσοχή σε μία αντίφαση, κύριε Επίτροπε. Κύριε Κατάινεν, εσείς τι μας είπατε ότι στην πολιτική συνοχής και στην ε, διαρθρωτική πολιτική ε, δεν ε, επιτρέπεται να πειραχθεί τίποτα να θίγει. Έχω ακούσει όμως και άλλες δηλώσεις και διάβασα και στη Λευκή Βίβλο του κυρίου Γιούνκερ με τα διάφορα σενάρια, στο σενάριο 4 αναφέρεται ακριβώς κάτι τέτοιο για την πολιτική συνοχή και την ορθωτική πολιτική που ανέφερε και η κυρία Κρέλ μπορεί όντω να διακυβευτεί για να βρούνε χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ. Και φυσικά με τρομάζει κάτι τέτοιο. Και μια ε, συνέντευξη της Επιτρόπου της κυρίας Γιούροβα που είπε ότι η πολιτική συνοχής ενδεχομένως στην επόμενη προγραμματική περίοδο να έχει καταργηθεί τελείως. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κάθε πολίτη στην Ευρώπη που περιμένει προστιθέμενη αξία από την Ευρώπη ακριβώς με τη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχή θα πρέπει να την γνωρίζει ή την έχει ήδη ζήσει. Και πραγματικά αυτά είναι φωνικά όπλα ε, ε, για να καταστρέψουμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Υπάρχουν αρκετέ πόλεις, μια που είμαι αρμόδια για το θεματολόγιο το αστικό, υπάρχουν αρκετέ πόλεις που δεν έχουν την παραμικρή δυνατότητα, όχι μόνο μικρές και μεσαίες, να φτάσουν σε χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ. Και θα πρέπει να τα πούμε όλα αυτά ξεκάθαρα και να φροντίσουμε να γράφονται και στις εκθέσεις και στις τροπολογίες μας αυτές τις ανησυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να θυμόμαστε όλοι το εξής. Μας λείπουν επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώς γι' αυτό δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Χρηματοδότηση όμως έχουμε. Στην αρχή όταν ιδρύθηκε το ΕΦΣΥ είπαμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τις πηγές χρηματοδότησης. Είναι πολλές οι πηγές. Αυτό που μας λείπει είναι έτοιμα έργα, όριμα προς εκτέλεση. Θέλουμε να δρομολογήσουμε λοιπόν έργα, γιατί αυτό μας λείπει. Και τι κάνουμε εμείς όλη αυτή την περίοδο για να έχουμε καλά έργα και να τα δρομολογήσουμε. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθούμε απλώς να ξεκλέβουμε διάφορα έργα που είναι όριμα προς χρηματοδότηση για να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές. Αυτά ακούω, ας πούμε, κάποια έργα που προετοιμάστηκαν για την πολιτική συνοχή ξαφνικά χρηματοδοτούνται από το τομείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Τι είναι αυτά εμείς θα πρέπει να δούμε πώς επεξεργαζόμαστε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια από τα κράτη-μέλη και πώς τα υλοποιούμε. Για να δούμε ποια είναι όριμα προς χρηματοδότηση και εκτέλεση και τι θα πρέπει να χρηματοδοτείται από ποια πηγή. Και από εκεί και πέρα να βρούμε τις συνέργειες που λέτε για να μην χρηματοδοτούμε τα ίδια έργα από διάφορες πηγές, αλλά να χρηματοδοτούμε διάφορες φάσεις ενός έργου από διάφορες πηγές και έτσι πραγματικά να βοηθούμε για την οικονομία μας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε που ήρθατε να μιλήσουμε στην Επιτροπή μας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Εγώ είμαι Ρουμάνος. Και θυμάστε ότι στη Ρουμανία υπάρχουν δυσκολίες. Την περασμένη εβδομάδα Ε, ήμουν σε ένα αεροπλάνο που πήγαινε από το Βουκουρέστι στο Κλους ε, και συνάντησα έναν ε, διοικητή τράπεζας και όταν του είπα γιατί δεν αξιοποιείς το σχέδιο Juncker, μου λέει τι είναι αυτό το πράγμα που μου λες. Κοιτάξτε, πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες στη Ρουμανία αγνοούσε τελείως την ύπαρξη του σχεδίου Juncker. Υπάρχει ε, ε, πρόβλημα με το σχέδιο Juncker. Ε, ε υπάρχει και εθνική διάσταση, αλλά είναι δυνατόν να αγνοούν οι μεγαλύτερες τράπεζες σε μια χώρα το σχέδιο Juncker. Δεν είχε ιδέα περί τίνος πρόκειτο, γιατί είναι αυτό το ταμείο. Υπάρχουν και άλλα ιδιωτικά ταμεία που περιμένουν χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό να λύθει αυτό το πρόβλημα. Και άλλη ερώτηση έχω που έχει σχέση με την πρόσβαση ε, στα ταμεία. Θα πρέπει να απλουστευτεί η διαδικασία. Όχι από τις Βρυξέλλες, αλλά δεν ξέρω, κάπως πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Να μην παραπέμπουμε τα πάντα σε κρατικό επίπεδο ενώ στην κεντρική κυβέρνηση. Υπάρχει εκεί η περιφερειακή αυτοδίκηση. Εγώ είμαι από το Κλούζ άλλο το Κλούς, άλλο, άλλο ε, το Βουκουρέστι. Είχαμε ένα σχέδιο επιχειρησιακό, ρυθμιστικό για το Κλούς. Ε, χρειαζόταν έγκριση των Βρυξελών, χρειάζονταν διάφορες διαδικασίες. Δεν είναι πάντα εύκολη η χρηματοδότηση. Πρέπει πάντα να περνάς από την κεντρική κυβέρνηση. Ξέρετε πώς έχουν αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο εύκολο στην απορρόφηση. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Στη Ρουμανία αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουμε καλές διαχειριστικές αρχές για να διαχείριζονται αυτά τα προγράμματα. Και έχω έρθει σε επαφή με τους διαφόρους ε, προσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Βρυξέλλες και έχω ρωτήσει τι γίνεται και τι γίνεται με τους Ρουμάνους για τις διαχειριστικές αρχές, γιατί δεν αντιγράφουν το πολωνικό μοντέλο, ας πούμε, που είναι βελτιστή πρακτική. Γιατί μου είπαν ότι α, είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία της κεντρικής ε, διοίκησης της κυβέρνησης στη Ρουμανία και δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πράγματα αποκεντρωμένα. Παρακαλώ κύριε Αντιπρόεδρε, ζούμε δύσκολους καιρούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να λύνουμε τα προβλήματά μας, τα προβλήματα και των κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να έχουμε μια πλουστευμένη διαδικασία για να μπορούμε να προχωρούμε. Σα είπα, στην Πολωνία αυτό το έχουν λύσει. Και στη Γερμανία, στη Γαλλία. Γιατί αλλού είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να δανειστούμε τις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών μελών. Ε, απλούστευση, εναρμόνιση και προβολή. Αυτό χρειάζεται. Δεν επιτρέπεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις το 34% των Ευρωπαίων πολιτών να γνωρίζουν τα θετικά της συμμετοχής της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το 34%. Φανταστείτε πόσοι αγνοούν τα ευρωπαϊκά ταμεία και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η Ευρώπη θα πρέπει να επικρατεί παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη γνωρίζουν οι πολίτες. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε. Υπάρχουν πολίτες που κατάγονται από χώρες καθαρού συνεισφορής. Ωραία. Και κοιτάνε και την πολιτική συνοχή και προβληματίζονται. Αλλά χωρίς την πολιτική συνοχή δεν νοείται Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τις περιφέρειες και την απομακρυσμένη περιφέρεια και να είναι εκεί ορατή και προβεβλημένη η περιφερειακή πολιτική και στις χώρες που είναι καθαροί συνεισφορεί. Γιατί βγαίνουν οι πολίτε και ρωτάνε πού πηγαίνουν τα λεφτά μου. Στην Ανατολική Ευρώπη. Ωραία. Σε ποιον, ποιο είναι ο τελικό δικαιούχο. Για να δουν ότι επανέρχονται με κάποιους μηχανισμούς στη δική τους εθνική οικονομία τα λεφτά αυτά, γιατί υπάρχουν πολλές εταιρείε από τη Δυτική Ευρώπη που εργάζονται στην Ανατολική Ευρώπη, ότι αυξάνεται το βιωτικό τους επίπεδο κτλ. Μου είπε ένα συνάδελφο από την Πολωνία ότι κάνανε επενδύσεις με τα διάφορα ταμεία και την πολιτική συνοχής. Έχτισαν ένα νοσοκομείο και το εξόπλισαν. Αλλά ποιος ε, παράγει τις συσκευές, η Siemens. Ε, τα λεφτά επιστρέφουν στους δωρητές. Ε, δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα <clears throat> ξεκομμένα. Υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές διαφορές ε, οι οποίες μειώνονται, κλείνει η ψαλίδα και αυτό είναι καλό και για τις χώρες που δίνουν τα χρήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νέλσον. Eh, eh, man κύριε lätt i diskussionen om nationella management system. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση για τα διάφορα συστήματα τα διαχειριστικά ίσως δεν είναι και η καταλληλότερη στιγμή να την κάνουμε. Πρέπει να δούμε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, έτσι ώστε να μην καταλήγουμε να χρηματοδοτείτε το ίδιο πρόγραμμα από δύο διαφορετικά ταμεία. Έχουμε διάφορα προβλήματα στη Σουηδία που έχουμε διαπιστώσει στον τομέα του συντονισμού στο, από τη πλευρά των εθνικών αρχών. Όταν εμπλέκονται περισσότερο του ενός ταμεία. Εάν, για παράδειγμα, πρέπει να ε, υπάρξει μια χρηματοδότηση και από ένα ταμείο γεωργική ανάπτυξης και από ένα ταμείο συνοχής ε, περιφερειακό ταμείο. Λοιπόν, όταν έχουμε ήδη τέτοιου τύπου προβλήματα, τι θα συμβεί όταν προσθέσουμε στο μείγμα ακόμα ένα ταμείο, το ΕΦΣΥ. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τις διάφορες εθνικές να, να αλλάξουν την προσέγγιση τους. Είπατε ότι θα χρειαστεί συνεργασία μεταξύ του ΕΦΣΥ και των περιφερειακών αρχών. Θα ήθελα να σας ζητήσω μήπως θα έπρεπε να επανεξετάσουμε και την αρχή της εταιρικής σχέσης, δηλαδή μήπως θα έπρεπε να κατά αναλογία να, να, να εφαρμόσουμε τον ίδιο κανόνα και να ζητάμε από τις εθνικές αρχές να συνεργάζονται με τις περιφερειακές αρχές. ως ένας τρόπος για να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση των χρημάτων του ΕΦΣΗ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το διαδικαστικό ερώτημα τώρα ή τουλάχιστον όχι, όχι σήμερα, μπορέσετε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για την παρουσία του εδώ στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική λειτουργία του Εύσεως τώρα. Έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη και έχει προωθήσει τις επενδύσεις. Στην εισαγωγική σας ομιλία μιλήσατε για την σημασία της γεωγραφικής ισορροπίας και για το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Γνωρίζω τις αρχές βάση των οποίων ε, αποφασίζονται, γίνονται, λαμβάνονται οι αποφάσει χρηματοδοτήσει από το ΕΦΣΕ δεδομένου ότι δεν πρόκειται για ένα ταμείο αλληλεγγύη ή για ένα ταμείο συνοχή. Όμω, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου, μόνο το 9% των κοντιλίων κατευθύνονται προς τα λεγόμενα νέα κρατημέλη, ενώ το 91% πηγαίνει προς τα 15 κρατημέλη πρώτου 2004. Προφανώς βέβαια άλλα ταμεία μπορεί να βοηθούν περισσότερο τα νέα κράτη-μέλη από ότι τα παλαιότερα. Όμως το ερώτημά μου είναι πώς μπορείτε να βοηθήσετε εκείνα τα μικρότερα κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα η Ρουμανία, που δεν καταφέρνουν να υποβάλουν στο ΕΦΣΙ ε, άρτια προγράμματα. Ο κύριος Φανίλστερ, ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Καθυστέρησα και δεν άκουσα την εισαγωγή του Αντιπροέδρου και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Μία ερώτηση έχω ουσιαστικά. Όπως είπε ο κύριος Κρέλ, η κυρία Κρέλ, συγγνώμη, υπάρχει κάποια επιφύλαξη ε, να επιστρέφονται πόροι από τα ταμεία αυτά στα κεντρικές κυβερνήσεις και μετά να επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με διάφορες αλχημίες να ξαναγυρνάνε στα κράτη-μέλη. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες τροπολογίες. Ε, όπως είπε και ο κύριος Νίλσον, τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν. Ε, μέσα σε ένα κράτος έχει διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης που έχουν συμφωνίες μεταξύ τους και έχουν συμφωνίες με εμπορικούς εταίρους, με παραγωγικούς φορείς, η τοπική αυτοδίκηση κτλ. Εκεί θα πρέπει και μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία να ε, αξιοποιούνται τα κονδύλια αυτά και να μπορούν να συνδυάζονται με τα μέσα του ΕΦΣΙ. Αυτό προβλέπεται ήδη στον ισχύοντα κανονισμό. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά επιστρέφουν τα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μετά κάπου ρέουν στην Ευρώπη. Στην νομοθεσία Omnibus είπαμε ότι θέλουμε να κόψουμε αυτή τη ε, δυνατότητα συγκέντρωσης και επιστροφής των πόρων. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση και περιμένουμε τις απαντήσεις και τα σχόλιά σας κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς για το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Θα υπάρξει μια διαδικασία fast track και, ε, κοινοποίησης, ε, μια ταχεία λοιπόν διαδικασία όπου στις περιπτώσεις που συνδυάζονται οι πόροι από το ΕΦΣΙ και από το ΕΦΣΙΦ. Γιατί στα έργα ΕΦΣΙ δεν υπάρχει κίνδυνος ε, κρατικών ενισχύσεων γιατί εξορισμού πηγαίνουν εκεί που δεν μπορεί να ε, ε, χρηματοδοτήσει ο ιδιωτικός ε, τομέας. Σε άλλες περιπτώσεις όμως θα υπάρξει αυτή η διαδικασία fast track. Αυτή είναι η δική μας πρόθεση και ήδη λειτουργεί στην πράξη. Επίσης είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι τώρα συζητούμε για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Αν δείτε τον κανονισμό Omnibus όμως Πρόκειται για, τη, για την περίοδο 2018-19-20. Δεν προεξοφλεί ή προδικάζει ε, την οποιαδήποτε έκφαση για επόμενη ε, περίοδο, προγραμματική περίοδο ή επόμενο ε, προϋπολογισμό, πόσο μάλλον τη Λευκή Βίβλο, που είναι μόνο ενδεικτικές οι προτάσεις και απολύτως στα χέρια των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω αυτό να διασκεδάσει τις ανησυχίες και τους φόβους σας ως προς τις προθέσεις μας. Όταν συζητούμε για συνδυασμό των πόρων ΕΣΥΦ και έψη, Εμείς δεν επιβάλλουμε σε κανένα να κάνει τίποτα, ούτε πιέζουμε να έχει συνδυασμό της χρηματοδότησης καθόλου. Εκείνοι όμως που είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιούν το έψη μαζί με πόρους ΕΣΥΦ θα κάνουν οικονομίες από τα ΕΣΥΦ για άλλους σκοπούς. Δηλαδή, the best αν θέλει κανείς να αξιοποιήσει όσο γίνεται καλύτερα τους πόρους που έχουν δοθεί στην περιφέρεια, με συνδυασμό, όσο περισσότερο συνδυάζεται το ΕΣΥΦ με το ΕΦΣΥ, Αυτός είναι ο μόνος λόγος λοιπόν συνδυασμού διαρθρωτικών ταμείων με ταμεία στρατηγικών επενδύσεων. για τις πόλεις και τις περιφέρειες και καμιά φορά και οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να συνδυάζουν διάφορες πηγές. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είναι καθόλου δεσμευτικό, είναι απολύτως προαιρετικό. Αν δεν θέλει μια περιφέρεια να το κάνει, δεν την υποχρεώνουμε, απλώς μειώνουμε την γραφειοκρατία και ε, διευκολύνουμε όσο γίνεται τη ζωή τους. Για τη συνοχή, η κυρία Κρέλ ρώτησε κάτι. Έχουν διαφορετικούς στόχους το Ταμείο Συνοχής και το, το ΕΦΣΙ και τα διαφορετικά ταμεία. Το ΕΦΣΙ σε χρηματοδότηση κάποια νοσοκομεία στην Πολωνία και κάποια πρωτοβάθμια κέντρα υγείας στην Ιρλανδία. Άρα υπάρχει μια μόχλευση ε, και βοήθεια στην ανάπτυξη των περιφερειών και των χωρών αυτό. Επίσης θα ήθελα να σας εξηγήσω ένα παράδειγμα που ακόμα δεν καταφέραμε να περάσουμε. Αυτό είναι μια ευκαιρία που υπάρχει στην Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε μεγάλους περιορισμούς οι ελληνικέ τράπεζε να αυξήσουν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μία από τις δυνατότητες θα ήταν να έχουμε πλατφόρμα χρηματοδότηση μικρομεσαίων με χρήματα ε, από τα διευθυντικά ταμεία, ε, κεφάλαιο και από, την, από το ΕΦΣΥ με κάποιες ιδιωτικές εταιρείε και να υπάρξει μια συγκέντρωση κεφαλαίου για να δανειοδοτεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό θα μπορούσε να είναι ο τρόπος να παρακαμφθεί η δυσκολία και τα προβλήματα που έχουν στην Ελλάδα οι τράπεζες αυτό τον καιρό. Και τώρα τα διαρθωτικά ταμεία θα μπορούσαν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά όπως σας είπα δεν καταφέραμε να πείσουμε ακόμα, ε, να, να στήσουμε αυτό το μηχανισμό στην Ελλάδα. Έχουμε πάντως ενθαρρύνει, παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να το κοιτάξουν. Τεχνική βοήθεια. Είναι και αυτή πολύ σημαντική γιατί έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε βελτίωση της γεωγραφικής κατανομής και μεταξύ κρατών μελών και εντός κάθε κράτους μέλους. Γι' αυτό το λόγο όλες αυτές οι προτάσεις για την ε, αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας είναι πολύ σημαντικές. Για ορισμένα έργα υποδομών χρειάζεται χρηματοδότηση με επιχορηγήσεις. Και εκεί μπορεί να υπάρξει συνδυασμός του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων με διαρθρωτικά ταμεία ή επενδυτικά ταμεία ή και άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το έύση για το τμήμα του χρηματοδότησης εκείνο που αφορά ιδιωτική επένδυση. Ε, με άλλα λόγια προσπαθούμε να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διάφορες ε, χρηματοδοτικέ πηγέ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. Όσον αφορά τον μελλοντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το Ηνωμένο Βασίλειο γνωρίζετε ότι δεν μπορώ να λάβω κάποια θέση ή να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον αυτή τη στιγμή. Είναι ένα από τα ανοιχτά ερωτήματα ε, στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν τα κράτη-μέλη, τα 27 και το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον όποια συμφωνία υπάρξει, εάν υπάρξει. κ. Σομερζή με ρώτησε εάν θα ήταν δυνατόν να δώσω κάποια στοιχεία φωτογραφικά αυτή τη στιγμή πώς είναι η κατάσταση ε, για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Το έχουμε ήδη πράξει αυτό αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ. Μπορείτε να βρείτε ε, στοιχεία, όχι τόσο αναλυτικά όσο θα ε, ήθελα, αλλά μπορείτε να δείτε πόσα χρήματα έχουν τευθυνθεί σε κάθε κράτος μέλος. Δεν πηγαίνει η ανάλυση σε βαθμό περιφερειών, αλλά έχετε για κάθε κράτος μέλος μια αναλυτική περιγραφή του ποιο ποσό έχει διαξιοποιηθεί. Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΦΣΥ, όλα τα προγράμματα, ε, στην ε, ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και με μια επεξήγηση πάντοτε της ε, δομής της χρηματοδότησης έχει εγκριθεί. Ορισμένε περιοχέ, ορισμένα κρατημέλη, ορισμένε εταιρείε έχουν ήδη αξιοποιήσει το ΕΦΣΙ και αυτό ίσω δώσει ιδέε ε, σε άλλε περιοχέ ή σε άλλε χώρε για το πώ θα μπορούσαν εκείνε να υποβάλουν προγράμματα και να το αξιοποιήσουν. κρατημέλη έχουν αξιοποιήσει περισσότερο το ΕΦΣΙ από ό,τι άλλα, βεβαίω. Ο λόγο είναι γιατί ε, σε αυτά τα κρατημέλη υπάρχει μια δημόσια αρχή η οποία προωθεί τη χρήση του ΕΦΣΥ και γιατί υπάρχει τεχνογνωσία οργάνωσης των, των προγραμμάτων και της υποβολής των προτάσεων. Αυτή η αρχή συνήθως απευθύνεται εκείνη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές εξηγώντας τους τι μπορεί να τους προσφέρει το ΕΦΣΥ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό ταξιδεύω συχνά σε πολλά κράτη-μέλη και προσωπικά το προωθώ το ΕΦΣΙ. Προσπαθώ να, το δημοσιο... την αξία του και να εξηγήσω σε τι μπορεί να συνεισφέρει μέσα από όλα τα κανάλια επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα. Αλλά είναι περιορισμένες οι δυνατότητες που μπορεί να έχει ένας Επίτροπο, η Επιτροπή συνολικά, εσύ ίσως ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ο καθένα εκλέγεται σε μια εκλογική περιφέρεια, έχετε καλύτερη επαφή με αυτές τις περιφέρειες και μπορείτε να το προωθήσετε πολύ καλύτερα. Το Τραμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ήταν μια πολύ σημαντική πηγή χρηματοδότηση για προγράμματα ενεργειακά στον τομέα τη ενέργεια και τη ενεργειακή υποδετικότητας. και ήταν ιδιαίτερο θετικό που διαπιστώσαμε ότι μέσω αυτών των προγραμμάτων μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε δια του ΕΦΣΥ νέε τεχνολογίε και καινοτομίε στον τομέα τη ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα από τη Δανία. Δημιουργήθηκε εκεί ένα ειδικό ταμείο από τα συνταξιοδοτικά ταμεία της Δανίας έχουν ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή τα συνταξιωτικά ταμεία της Δανίας γιατί ε, δεν έχουν αρκετά υψηλό ρυθμό απόδοσης ε, στις επενδύσεις που είχαν έως στιγμής. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουν σε ε, προϊόντα που τους φέρουν μεγαλύτερη απόδοση. Αλλά απ' την άλλη δεν θέλουν να λάβουν και μεγάλο ρίσκο. Άρα χρησιμοποιούν το EFC ως ένα μαξιλάρι ασφαλείας έτσι ώστε εάν το ε, συνταξιοδοτικό ταμείο υποθέσουμε ότι χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας το οποίο τελικά οδηγήσει σε ζημίες, δεν ε, δουλέψει, ε, η ζημία αυτή θα απορροφηθεί αρχικά μέσω του ΕΦΣΙ, γιατί η χρηματοδότηση έγινε μέσω του ΕΦΣΙ. Ζητήσατε επίσης να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για το ποιες είναι, ποιοι, είναι οι τελικοί δικαιούχοι ε, που έχουν υποφεληθεί από το EFSI και πόσοι από αυτούς είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προβλέπουμε ότι περίπου 100.000 400.000 ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υποφεληθούν εν καιρό. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη αξιοποιήσει τα χρήματα που τους έδωσε η e FSI. Χρήσιμο επίσης θα ήταν όταν μια μικρομεσαία επιχείρηση αξιοποιεί τα χρήματα αυτά να φτάνουν τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, γιατί μερικέ φορέ η χρηματοδότηση γίνεται μέσω μια τράπεζα και η τράπεζα δεν λέει αναγκαστικά στον πελάτη τη ότι η χρηματοδότηση που του παρέχει είναι εφικτή επειδή υπάρχει μια βοήθεια από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση θα αυξήσουμε τη χρηματοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του EFSI. Ε, Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη τη Επιτροπή σα για αυτή τη συζήτηση. θεωρώ πολύ σημαντική και α ε, παραμείνουμε. Όπω ζητώ συγγνώμη. Κάτι ξέχασα να απαντήσω. Κανονικά δεν Δεν μου συμβαίνει ποτέ, αλλά. Το ερώτημα του κύριου Φανίλ θα το βρω τώρα αμέσω. Yes. Um, if I Ναι, λοιπόν, αν σωστά αντιλήφθη το ερώτημά σα, Ε, δεν υπάρχει κίνδυνος τα χρήματα να γυρίσουν πίσω. Δηλαδή, ε, εάν κανείς συνδυάσει χρηματοδότηση διαφθρωτικού και επενδυτικού ταμείου αφενό και ε, και Δεν υπάρχει ο κίνδυνο χρήματα που πήγαν, κονδύλια που έφτασαν σε μια περιφέρεια να γυρίσουν πίσω στι Βρυξέλλε. Δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Ε, αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια περιφέρεια η οποία θέλει να υποβάλει ένα πρόγραμμα και να ζητήσει χρηματοδότηση και από τα δύο ειδών ταμεία, σημαίνει ότι έχει λάβει την απόφαση συνειδητά. Τα διαρθρωτικά ταμεία βρίσκονται στα δικά τους ε, χέρια η χρηματοδότηση και από το Διαρθρωτικό Ταμείο και από το ΕΦΣΙ θα φτάσει στην περιφέρεια, εάν τελικά υλοποιηθεί το πρόγραμμα φυσικά. Εάν από την άλλη η επένδυση δεν γίνει, δεν πρόκειται να γυρίσουν χρήματα ούτε στις Βρυξέλλες ούτε στο Λουξεμβούργο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του ΕΦΣΙ και του συνήθου τρόπου με Αναφερόμαστε στο άρθρο 125 του Omnibus, αλλά χαίρομαι για την απάντηση που μου δίνετε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Βοηθά αυτό. Είναι κάτι χειροπιαστό το οποίο μπορούμε να μεταδώσουμε, γιατί θυμάμαι ότι στις πρώτες συζητήσεις που είχαμε για το FC, ε, είχε ελεγχθεί ότι θα ξεκινήσουμε με κεντρικώς ε, συντονιζόμενα προγράμματα στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020, και τώρα πια βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτή η διαδικασία χωρίς να περιμένουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο του, του, του, του προπολογισμού. Ε, και θα μπορούσαμε να τη διευκρινίσουμε αυτή τη διαδικασία μάλλον αυτή τη στιγμή αξιοποιώντας τη, τη, τη συζήτηση για το Omnibus μέσω τροπολογιών, αν συμφωνείτε και εσείς. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για τις απαντήσεις που δώσατε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τη συζήτηση, ιδιαίτερα για αυτή την τελευταία απάντηση που δώσατε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δείχνει και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, πώς να κινηθεί στο θέμα της συζήτησης για το Omnibus. Σας ευχαριστώ. Πριν από έναν χρόνο είχατε έρθει το Μάιο του 2016 ε, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ελπίζω να μην περάσουν πάλι 12 μήνες μέχρι να σας ξαναδούμε. Ελπίζω, ελπίζω. Θα δούμε πάντοτε είναι χαρά για μας να σας υποδεχόμαστε εδώ και να συζητούμε τα διάφορα προβλήματα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Okay. Thank you very much. Okay, on this point I close, uh, Λοιπόν, αυτή ήταν η δημόσια συνεδρίασή μας. Ακολουθούν οι συντονιστές και κλεισμένων των θυρών και παρακαλώ όλα τα μέλη που δεν είναι συντονιστές να αποχωρήσουν τις αιθούσεις. Ευχαριστώ. Θυμίζω ότι αύριο το πρωί έχουμε ψηφοφορίες, στις 8.30 ώρα αρχίζουμε, και όχι 9. Ψηφοφορία 8.30 ώρα ακριβώς.